νομοθεσία. Επίσης υπάρχει μια πρόταση για τον Γιώχαν Κορνέλιους Ντεν ε, ως ε, μέλους της Επιτροπής για τη Συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκθέσω τον κύριο Πλάνη, ρωτώ αν υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτό. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν αυτή η θέση και με βάση το άρθρο 3, παραγράφων 3 και 4 του κανονισμού θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στη συνεδρίαση 22 Μαρτίου του 2010 επιβεβαίωσε την ε, εντολή της κυρίας Λουγκρίπ και του κυρίου Κοσμόφσκι και παρακαλώ να επικαιρώσει το σώμα την εντολή αυτή, τις εντολές αυτές. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Επομένως επικυρώνονται οι εντολές των ε, οι βουλευτικές θέσεις των δύο αυτών συναδέλφων. Τώρα περνούμε στις, ε, στα νομοθετήματα που εξετάζονται με τη διαδικασία της συναπόφασης. Θα σας ενημερώσω ότι συζητήσαμε